δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τη Λευκορωσία. Ω συνήθω, θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Κύριε Υφυπουργέ Βόντρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να θέσουμε στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου το ζήτημα αυτό. Να ξεκινήσω εδώ με μια θετική νότα. Παρατηρήσαμε με ικανοποίηση τα διαβήματα που ανέλαβε η Λευκορωσία τις τελευταίες εβδομάδες ειδικά σε ό,τι φορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την διανομή εφημερίδων όπως η Ραντόνια Νόβολατ ή το Νάσια Νίβα. Επίσης, επίσης ρύθμιση για το διαδίκτυο και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Ξεκίνησαν επίσης διαβουλεύσεις με τον ΩΣΑ για τη βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας. Αυτά τα βήματα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση των κριτηρίων που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, προϋπόθεση για την ε, διατήρηση της ε, βίζας για περίοδο πάνω των 6 μηνών. Αυτό τον. και αυτό χάρη σε επαφές που είχαμε με τη διοίκηση της Λευκορωσίας. Πρέπει να λάβουμε απόφαση όμως στις αρχές Απριλίου. Θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε τις πολιτικές επαφές σε διμερές επίπεδο και όχι μόνο για να εθαρρύνουμε την Λευκορωσία να προχωρήσει προς την οδό που χαράξαμε. Και αυτό αναφέρεται συμπέρασματα του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου Ως ε, μήνυμα ενθάρρυνσης η Προεδρία μας προτίθεται να οργανώσει μια άλλη διυπουργική τρόικα με τη Λευκορωσία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις της ελευθερίας στην χώρα δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Συζητάμε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Ο κύριος Μπάρι και άλλοι αντικαθεστωτικοί με τους οποίους συζητάμε όπως ο Αλεξάνδρου Μπιλίνκεβιτς, ο κ. Σκόζουλιν αλλά και άλλοι. Η Λευκορωσία όσο γνωρίζετε είναι μία από, ένα από τα έξι κράτη με τα οποία έχουμε αναπτύξει σχέσεις στο πλαίσιο της ανατολικής της γειτονίας προτιθέμεθα να προαγούμε αυτήν την ε, συμφωνία γειτονίας ε, τον Μάιο στην Πράγα θεωρούμε ότι μέχρι τώρα θα έχει περάσει εξαμήνως ε, περίοδος και θα μπορούμε να κάνουμε την απαραίτητη αξιολόγηση. Πιστεύουμε πως ε, χρειάζεται ε, να υπάρξει επικοδομητική στάση από πλευρά Λευκορωσίας. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην θεωρούμε ότι θα υπάρξουν τεράστιες αλλαγές ο Λουκασέγκο ε, προσπαθεί να διατηρήσει πολύ στενές σχέσεις ε, με την Μόσχα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμεί έχουμε κάποιε αρχέ. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προ τον Λουκασέκο και να χρησιμοποιήσουμε τι ευκαιρίε που μα ε, παρέχονται για να ενθαρρύνουμε μια δυναμική η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο θα ξεκινήσει στην Λευκορωσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να μιλώ για την Λευκορωσία, γιατί σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι και χαρήκαμε που το διαπιστώσαμε αυτό. Η Λευκορωσία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, όχι επειδή είναι μόνο επειδή είναι μια χώρα που χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση της περιοχής. Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία. Βρισκόμαστε, αν θέλετε, εν το μέσο, στο μέσο το, της αναστολής των έξι μηνών για την απαγόρευση θεώρησης ε, των αξιωματούχων της Λευκορωσίας. Όταν ε, θα λήξει αυτή η αναστολή στις 30 Απριλίου. Τώρα είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για το αν οδεύει προς σωστή κατεύθυνση η Λευκορωσία. Για το κατά πόσον θα συνεχιστεί κιόλα η αναστολή αυτή και θα αναλυφθούν σωστά μέτρα. Η θετική πρόοδος που ξεκίνησε με την απελευθέρωση των ε, εναπομείναντων πολιτικών κρατουμένων θα πρέπει να συνεχιστεί για να συνεχιστεί και η αναστολή της απαγόρευσης. Θα θέλουμε συγκεκριμένη πρόοδο να μην γίνουν άλλες πολιτικές κρατήσεις, συνεργασία με τον ΟΑΣΥ, με το ΟΔΙΡ για τις μεταρρυθμίσεις της εκλογικής νομοθεσίας, ελευθερία του τύπου, καλύτερες συνθήκες λειτουργίας για τις ΜΚΟ και να μην υπάρχουν πολιτικές κρατήσεις και επίσης να υποστηριχθεί η ελευθερία του θα πρέπει να πω ότι σημειώθηκε πρόοδος στους τελευταίες τρεις μήνες, για παράδειγμα σε διαφορά την άρση της απαγόρευσης δύο μεγάλων εφημερίδων, οι οποίες πλέον ελεύθερα κυκλοφορούν. Κατά δεύτερον, η οργάνωση του κυρίου Μιλικέβιτς για την ελευθερία, η οποία μπόρεσε να καταχωριστεί τελικά. Και τρίτον, διαβουλεύσεις μεταξύ ε, Οντύρ και Λευκορωσίας για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Αυτή η πρόοδος ήταν η άμεση αντίδραση των ετοιμάτων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Νοεμβρίου και μας ενθαρρύνουν. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή στις σχέσεις μας και αν θέλουμε να συνεχιστεί και η αναστολή της απαγόρευσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο στην ελευθερία του τύπου και για το διαδίκτυο και για την διαπίστευση των ξένων δημοσιογράφων. Επίσης, θα πρέπει να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες καταχώρησης και για τις συνθήκες λειτουργίας των ΜΚΟ και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα του κ. Μπαραζένσκα, των ακτιβιστών. Και θα πρέπει να δούμε αποδείξεις ότι υπάρχει περιθώριο για φιλιρινικές διαμαρτυρίες. Η πρόοδος, ωστόσο κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι το αμφίδρομο και αν η Λευκορωσία μπορεί να σημειώσει αυτή τη σημαντική πρόοδο, νομίζω ότι είναι εξίσου απαραίτητο να είμαστε κι εμείς ε, να απαντήσουμε με σημαντικό πακέτο μέτρων. Έχει καταρτήσει κάποιες ε, προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμπεριλάμβαναν τα εξής επέκταση του τεχνικού διαλόγου που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο για τον ενέργεια και το περιβάλλον και σε άλλους τομείς, μια συμβολική αύξηση αν θέλετε των κονδυλίων για την Λευκορωσία για να υποστηριχθούν οι συζητήσεις αυτές και ενίσχυση της Λευκορωσίας να προσαρμοστεί, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει. Και τέλος, να εντατικοποιηθούν στις 26 Ιανουαρίου όταν η Τρόικα θα συναντηθεί με τον, με τον πρόεδρο εξωτερικών Μάρτινοφ και όπου σκοπεύω να πω με σαφήνεια στο Μάρτιν τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελευκορωσία, να κάνουμε και εμείς μία πρόταση όμως και φυσικά η εντατικοποίηση του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στις συναντήσεις των βουλευτών στο Μίνσκ, για παράδειγμα με βουλευτές ε, της Λευκορωσίας, γιατί όχι, ένα άλλο θέμα θα ήταν η δυνατότητα ε, ανοίγματος συζήτησης για θέματα διευκόλυνσης βίζας. Γι' αυτό λοιπόν το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Συμβουλίου και είναι σαφές ότι θα πρέπει να σημειωθεί και περαιτέρω πρόεδρος από τη Λευκορωσία, αλλά θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον φυσικά αναγνωρίσουμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Τέλος, Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε το πλήρες δυναμικό του ENP και της ε, Ανατολικής εταιρικής Σχέσης για να βοηθήσουμε την Λευκορωσία και σε ό,τι αφορά το PCA και την αύξηση της ενισχύσης μας μετά τις 30 Απριλίου, αν κριθεί ότι έχει σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος, θα δούμε αν θα συνεχιστεί η αναστολή της απαγόρευση, αν είναι αρκετή η πρόοδος της Λευκορωσίας, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε κι εμείς και ελπίζω πραγματικά να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο με τη Λευκορωσία. Thank you very much. We start our debate. Uh, Ευχαριστώ. Πρώτος αγορτής ο κύριος Προτασίβιτς ε, από πλευρά ΣΕΛΚ, ο οποίος και προεδρεύει της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λευκορωσίας. Παρακαλώ για, λεπτά, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ Βόντρα. Ο λόγος για τον οποίο ε, συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο στη μέσα διάταξη των εργασιών μας είναι πως ε, ε υπάρχει έχει περάσει ικανή περίοδος ε, από την κατάρρηση απαγόρευση πολιτικών επαφών με λευκορωσικέ αρχέ και αστολή τη απαγόρευση θεώρηση ε, για του αξιωματούχου Θεωρούμε λοιπόν ότι το κίνημα του Μιλινκέβιτ ε, αποκαταστάθηκε και επίση ε, δύο εφημερίδε ξανακυκλοφορούν ελεύθερα. Πρέπει να το καταδικάσουμε το γεγονό ότι η πολιτική ε, κρατούμενοι, οι οποίοι ελευθερώθηκαν να πρεθούν την περασμένο χρόνο, δεν ε, χαίρουν όλων των ε, πολιτικών τους ε, και άλλων δικαιωμάτων ε, για να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ελευθεροτυπία και να τεθούν σε εφαρμογή τα άρθρα του ποινικού κώδικα τα οποία είχαν καταργηθεί. Μάλλον θα πρέπει να καταργηθούν κάποια άρθρα όπως το 193, 367, 368 και 369 του ποινικού κώδικα. Στο ψήφισμα που συζητάμε σήμερα, ζητάμε από την Λευκορωσία να μην περιορίσει τις δραστηριότητες μη κυβερνικών οργανώσεων ή των μέσων επικοινωνίας. Πρόκειται για μια έκκληση η οποία πάει προς δύο κατευθύνσεις ε, συνάμα, διότι απευθύνεται και προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν, διότι θα πρέπει να ε, πάψει την χορήγηση θεωρήσεων ε, εάν ε, η Λευκορωσία δεν συμμορφωθεί. Επίσης επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας ε, προκειμένου να ε, χορηγηθούν τα κονδύλια που είναι απαραίτητα προς τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής ο κύριος ε, Παλέκης, ε, του των Σοσιαλιστικής Ομάδας, για δύο λεπτά. Τρία λεπτά, τρία λεπτά, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κύριε Φιμπουργέ, υπάρχει μία παλιά αγγλική παρεμία ότι όσο πιο ψηλή είναι τα σύνορα μεταξύ των γειτόνων, τόσο καλύτερες είναι οι σχέσεις τους. Εμείς θα πρέπει να χαμηλώσουμε, αν θέλετε, τους φράχτες που μας χωρίζουν σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα. Λόγω των αυταρχικών του τάσεως, η Λευκορωσία έγινε, αν θέλετε, ο άρρωστος της Ευρώπης. Η χώρα απομονώθηκε έχασε και την έδρα της στο Συμβούλιο της Ευρώπης πέρυσι η ελπίδα για την ε, αναπτέρωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναγεννήθηκε. Έγιναν κάποια μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση από τις αρχές της Λευκορωσίας σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους, τη δημοσίευση ανεξάρτητου των εφημερίδων και θυμόμαστε επίσης και την ε, σχετική ευρωπαϊκή αποστολή. Νομίζω ότι ο ουρανός σιγά σιγά καθαρίζει παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες ενώπιον μας. Ο κ. Προστατσέβης σωστά ανέφερε ποια είναι αυτά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η χώρα βρίσκεται το χείλος ε, σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ζωής του καθημερινού ανθρώπου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί την οδό της αμοιβαίας κατανόησης. Καταρχάς θα πρέπει θα πρέπει να καταργήσουμε την οικονομική επιβάρυνση για την χορήγηση θεωρήσεων προς τους πολίτες της Λευκορωσίας αναφορικά με τα πρινικά εργοστάσια της Λευκορωσίας. Θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο αυτό όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στο Βίλνιους. Και άλλες χώρες προγραμματίζουν την κατασκευή τέτοιων εργοστασίων. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί λοιπόν ο διάλογος μεταξύ των χωρών αυτών. Και οι Βρυξέλλες θα πρέπει να συνεχίσουν να επιβλέπουν κατά πόσο τηρούνται οι συστάσεις της Διεθνής Επιτροπής, της Επιτροπής για την Ατομική Ενέργεια. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε πρόοδο στην Λευκορωσία αν δεν πέσουν, αν θέλετε, τα όρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας. Θα πρέπει να συζητήσει η κυβέρνηση και με τους εκπροσώπους των ε, οργανώσεων της νεολαίας. Σε κάποιους ε, μήνες, αντί τρεις μήνες, θα συζητηθεί κατά πόσο θα συνεχιστεί η αναστολή. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, από το φιλελεύθερους, ο κ. Σονισκεβίτς, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Από τη Λευκορωσία λαμβάνουμε κάποια μηνύματα τα οποία είναι διφορούμενα. Βλέπουμε αφενός ε, την απελευθέρωση πολικών κρατουμένων, αλλά και από την άλλη πλευρά απαγόρευση κάποιων κινημάτων. Αλλά έχουμε και άλλες συλλήψεις αντικαθεστωτικών και περιορισμό για καταπάντηση των ελευθεριών Παράλληλα υπάρχουν πολλές κειμενικές οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην λειτουργία τους. Σε ορισμένες περιπτώσει εφαρμόζεται και η θανατική ποινή. Εμεί δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στην χώρα αυτή. Θα πρέπει να εγγυθούμε το διάλογο ανάμεσα στου εκπροσώπους του Κοινοβουλίου μας και του εκπροσώπου τη Λευκορωσικής Βουλής και σε αυτό αναφέρεται και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται λοιπόν να μειώσουμε το κόστος για την έκδοση των προξενικών θεωρήσεων για τους πολίτες Λευκορωσίας. Αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικέ επιπτώσει σε όσους επιθυμούν να ε, εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται παράλληλα να βοηθήσουμε και οικονομικά την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Ε, πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτων οργανώσεων και τον ε, τύπο. Στην Ευκορωσία ο μοναδικός ε, βασικός εργοδότης είναι το κράτος, το οποίο όμως αυτό που κάνει είναι να χορηγεί αιτήσεις συμβάσεις στους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια εμείς θέλουμε να προσεγγίσει η χώρα αυτή τα ευρωπαϊκά στάνταρ και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα σε εμά και τις λευκορωσικές αρχές. Ο κύριος Τσέρνες και έχει το λόγο ο της ΟΕΝ για 1,5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσβάτως ε, συζητήσαμε για το πρόβλημα της Λευκορωσίας. Αυτό αποτελεί έναν τρόπο εποπτείας των όσων εξελίσσονται στην χώρα αυτή, η οποία είναι και η γειτονική μας. Η διαδικασία ε, δημοκρατισμού στην Λευκορωσία είναι ικανοποιητική. Όχι. Υπάρχουν εκατοντάδες λόγοι για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Εμεί όμως την πλάτη δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε στη χώρα αυτή. Μπορούμε να μιλήσουμε για ελευθεροτυπία, για δημοκρατία, για ελευθερία κλπ. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να ρίξουμε κόκκινη κάρτα στην ε, Λευκορωσία για πολλά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι Λευκορώσοι είναι Ευρωπαίοι. Και ο πολιτισμός της Λευκορωσίας είναι πολιτισμός της Ευρώπης. Στην ε, Λευκορωσία οι πολίτες αγωνίζονται για τις ελευθερίες τους, για την θρησκευτική ελευθερία κλπ. θα ήταν ε, πραγματικά απόλυτα ανεύθυνο από πλευράς μας ε, να μην δώσουμε σημασία στα τεκτονόμενα στην χώρα. Να, το να πρέπει να απαγορεύσουμε ο Λουκασέγκο να διώκει τους ε, χριστιανούς ε, ιερείς αλλά παράλληλα θα πρέπει να φροντίσουμε η Λευκορωσία να μην ε, ενταχθεί στην σφαίρα της Σοβιετικής Ένωσης. Ο κύριος Όρατσοκ έχει τον λόγο τώρα. Zdravím české předsednictví pod vedením θα ήθελα να καλωσορίσω την Τσεχική Προεδρία. για την ελευθέρωση των ε, πολιτικών κρατουμένων. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις θετικέ από πλευρά Λευκορωσίας. Θα πρέπει να δούμε τώρα αν πίσω από τη διάθεση για διάλογο υπάρχει πραγματική διάθεση για μεταρρύθμιση και ανα κλειτέρωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή η Λευκορωσία έχει θέση στην Ευρώπη και εδώ και πολύ καιρό περιμένουμε να ξαναρχίσουν οι σχέσεις μας, αλλά υπό σαφείς όρους και αυτό κυρίως περιλαμβάνει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης, αλλά για το σύνολο του πολιτικού και κοινωνικού οικοδομήματος. Η διαφθορά και η καταποίηση δεν είναι πράγματα που έχουμε ξεχάσει. Θα τα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε. Τον ε, Οκτώβριο αποφασίσαμε να ανασταλθεί η απαγόρευση ταξιδίου του Προέδρου Λουκασέγκου. Είναι σημαντικό να επιτραπούν και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στη Λευκορωσία για να καταστούν δυνατές οι συζητήσεις και με τους ε, αντικαθεστωτικούς, γιατί η εμπειρία μας διδάσκει ότι κάθε δικτατορία κάποια στιγμή τελειώνει. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από την ΚΟΕ, τον λόγο έχει η κυρία Φλασάρβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Λευκορωσία είναι η τελευταία χώρα με την οποία δεν έχει ειδικέ συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο. Αυτό θα μπορούσε να λάβει τέλος σύντομα. Η περίοδος δοκιμής θα λήξει σύντομα. Η Λευκορωσία μπορεί να έχει λίγο παραπάνω δημοκρατία και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει τους όρους για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Οι πρόσφατες αλλαγές πάντα γίνονταν στα πλαίσια του διεθνούς ε, συγκειμένου. Σήμερα μετά από τις δεκαετίες ε, της ισχύω της, ε, των ΗΠΑ βλέπουμε αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων. και αναζητώνται νέες ε, ισορροπίες. Η Μολδοβία, όπως και ο Κάφκασος, αποτελούν σημείο διένεξης πολλών παραγόντων. Θα ήταν παράλογο να το αρνηθούμε αυτό, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Οι πραγματικές αξίες εδώ πέρα είναι η στρατηγική, τα χρήματα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει για τη δημιουργία ενός διεθνούς, ε, νέου διεθνούς ε, πλαισίου. Ο κύριος ε, Φιόρε, ο κύριος Βέλτερ. Βέλτερ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόγνωση αυτή που ακούσαμε στην αρχή για τον πρόεδρο Λουκασέγκο στην αρχή του έτους βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπο με μια οικονομική κρίση και προϋπόθεση ήταν ε, στις 2 Ιανουαρίου η μείωση της αξίας του ρουβλίου που έπληξε τους πολίτες. Πλέον το ευρώ στο Μίνσκ είναι πολυπόθετο. Αυτή η απίσχναση της οικονομικής θέσης στη Λευκορωσία θα αλλάξει την στάση του Λουκασέγκο. Πέρα από τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα, πρόκειται για αισθητικέ αλλαγές του Λουκασέγκο. Ο πρόεδρος πολύ απλά θα προσωμείωνε μία προσέγγιση προς τη, στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες δυνάμεων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθεί με σαφείς πολιτικές σε αυτό το σενάριο. Όλα θα, τα, όλες οι αρχές της Λευκορωσίας θα πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σημαντικούς ε, στόχους. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Φιόρε. Δύο λεπτά. Ε, Πρόεδρε, νομίζω πως δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι ώστε να διατηρήσουμε η αδίποτε μορφή κύρωσης απέναντι στην Λευκορωσία. Εδώ βλέπουμε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει μια κρίση όπως και όλα οι χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για μια χώρα η οποία, η οποία η, είναι ελεύθερη. Πριν από μερικούς μήνες γνώριζε μια ανάπτυξη της τάξης του 80% και δεν εμποδίζει τους αλλοδαπούς, τους Ευρωπαίους να αγοράζουν οικόπεδα και κατοικίες στην χώρα αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σκεφτική ελευθερία, προ καιρού ο Καρδινάλιος Μπερτώνε μετέβη στην Λευκορωσία και φυσικά δημιουργήθηκαν σχέσεις ανάμεσα στο Βατικανό και την Λευκορωσία. Ε, συμφωνήσαμε σαν αναγνώρισης και σεβασμού. Μιλήσαμε για κάποιους ε, φυλακισμένους, μιλάμε για τρεις πολιτικούς ε, κρατούμενους οι οποίοι όμως απελευθερώθηκαν. Μιλάμε για πολιτικές εκλογές οι οποίες φυσικά δεν ε, είναι όμοιες ε, με τις ε, δικές μας εκλογές, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν δώσει και ώρα, ώρας εκπομπών στην τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Γνωρίζουμε ότι κάποιες εφημερίδες ανεξάρτητες αυτές τις εβδομάδες θα έχουν την δυνατότητα να διανέμονται. Πιστεύω ότι δεν είναι προς όφελος της Ευρώπης να ε, έρθει σε σύγκρουση με την Λευκορωσία, διότι η Λευκορωσία είναι μια πολύ σημαντική χώρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ρωσία. Έχει μια πολύ μεγάλη καθολική κοινότητα που κάνει την χώρα αυτή να είναι ένα στρατηγικός εταίρος, στρατηγικός σύμμαχος Πρόκειται για ένα παράδοξο σήμερα να μιλάμε για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, ενώ η Λευκορωσία ε, παίζει έναν ρόλο πολύ σημαντικότερο, πολύ πιο ενδιαφέρον ως εταίρος της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα εκ μέρους ε, του ΕΛΚ ο κύριος Ντούκα Ζόνονμι. Ευχαριστώ. Οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσία έχουν φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο. Είναι δύσκολο να αναλάβουμε δράση. Ακούσαμε διάφορα για τη Ρωσία, Λευκορωσία, για την διένεξη με την ε, και την παγκόσμια κρίση. Ο Λουκασέγκο αφήνει, απελευθερώνει κάποιους πολιτικούς ε, κρατούμενους, ε, αφήνει να δημοσιευτούν κάποιες εφημερίδες και όλα αυτά ε, αποτελούν, αν θέλετε, μόνο τα φαινόμενα στα πλαίσια μιας πραγματικής ε, προσέγγισης. Το Μίνσκ θα πρέπει να ανοίξει την πολιτική του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όντω να εξαντλήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Μπορεί να ασκήσει πίεση στην πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή και γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποια πολιτική ασκείται στις Βρυξέλλες και είναι σημαντικό για το σκοπό αυτό να εποπτεύουμε και να παρακολουθούμε τον, το πακέτο των συνθήκων και των όρων που έχουμε επιβάλει. Δεν είναι προφανές ούτε πιθανό να αλλάξει πραγματικά ο Λουκασέγκο. Θα πρέπει όντως να στηρίξουμε την αντιπολίτευση και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και στο εκλογικό σύστημα και στο ποινικό σύστημα για την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους. Γιατί οι χώρες της περιοχής αυτής έχουν καταδείξει ότι χωρίς ε, σαφείς όρους δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ, αν θέλετε, μια πραγματική δημοκρατική διαδικασία. Ο κύριος Πινιόρ, λέει ο πρόεδρος, για δυόμιση λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ, να υπογραμμίσω ως θετικό στοιχείο την παρουσία εδώ ανάμεσά μας του Υπουργού Βόντρα. Θεωρώ πως ε, αυτό καταδεικνύει ποιος είναι ο ρόλος που η Τσεχική Προεδρία αποδίδει στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναλύουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απέναντι στην ε, Λευκορωσία. Αναλύουμε μια στρατηγική ανοίγματο, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε εδώ και μερικούς μήνες. Ο απολογισμός αυτής της στρατηγικής, κατά την άποψή μας, είναι θετικός. Εξάλλου αυτό αναφέρεται και στο σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Στο Μίνσκ όντως ε, ιδρύθηκε η μόνιμη εμπισοπία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξάλλου λάβαμε κάποια θετικά μηνύματα αναφορικά με ζητήματα ελευθερίας όπως η καταχώρηση του κινήματος για την ελευθερία του Μιλικέβιτς στα Μητρώα επίσης ε, επιτράπηκε η ε, καταχώρηση δύο ανεξαρτήτων ε, εφημερίδων και έχω κατά νου επίσης και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Λευκορωσίας σχετικά με την ε, θετική αντιμετώπιση από πλευράς Λευκορωσίας ε, της ε, εταιρικής σχέσης. Οι αρχές Λευκορωσίας επίσης αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της αφχαζίας Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία που αναφίβολα οφείλονται και στην ευνοϊκή αντιμετώπιση της χώρας από τις Σοβιετική Φυσικά στο σχέδιο ψηφίσματος μιλάμε και για κάποιους περιορισμούς που ήδη υπάρχουν στην χώρα αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεν είναι μια ολοκληρωμένη δημοκρατία η χώρα αυτή. Έχω κατά νου αυτά τα οποία είπε η κυρία Βάλνερ. Αυτή η διακοπή των κυρώσεων θα καταστεί δυνατή μόνο όταν απελευθερωθεί η οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ε, μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της χώρας, Πρόεδρος. Θα ήθελα να παρατηρήσω πως ε, στις συζητήσεις αυτές πάντα παρίσταται εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετική περίπτωση. Ε, φυσικά εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία του Υπουργού Βόντρα. Δεν θέλω να αφαιρέσω τίποτα από την σημασία της ε, παρουσίας του. Κύριος Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, οι σχέσεις με την Λευκορωσία εξαρτώνται από δύο παράγοντε. Αν υπάρξει βούληση και από τι δύο πλευρέ, τότε θα υπάρξει διάλογος. Υπάρχει το θέμα της ε, γειτονία και της ε, Ευρωπαϊκή Εταιρική σχέση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δέχομαι με ικανοποίηση την πρόσφατη πρόταση τη ε, πρωτοβουλία μάλλον τη Κομισιόν για τη βελτίωση τη σχέση με την ε, Λευκορωσία. Να πω ότι η Λευκορωσία έκανε πολλά προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Παραδείγματο χάρη επέτρεψε την ε, ελεύθερη διανομή δύο εφημερίδων και την καταχώρηση του κινήματο για την ελευθερία στα Μητρώα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές προσδοκίες από πλευρά ε, της Λευκορωσίας σε πολλά θέματα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συμμετρία και αμοιβαία κατανόηση. Οι αρχές Λευκορωσίας θα πρέπει να θέσουν τέλος στην ε, ε, επιβολή κάποιων όρων για την έξοδο από την χώρα. Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθάει στην κατάσταση αυτή, δεν μειώνει το κόστος των θεωρήσεων και αυτό αφορά ιδιαίτερα τους, όσους κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές. Τώρα υπάρχει και το διακόπτη ο Πρόεδρος. Εξαντλήσατε το χρόνο σας, αυτό ισχύει για όλους. Ένα λεπτό είναι ένα λεπτό και όχι παραπάνω. Το λόγο έχει ο... η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για την ευρωπαϊκή πολιτική αναφορικά με τη Λευκορωσία, για τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να εστιαστώ σε ένα σημείο για την απαγόρευση ταξιδίων για τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δίνω προσοχή και στα υπόλοιπα θέματα που αναφέρθηκαν. Θα ξέρετε βέβαια ότι τα παιδιά, τα θύματα του Τσέρνομπιλ έρχονται στην Ολλανδία αλλά και σε, άλλε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνέλθουν λίγο μετά την καταστροφή αυτή. Μιλάμε για παιδιά τα οποία γεννήθηκαν μετά την καταστροφή, έχουν την ηλικία που είχα εγώ τότε όταν έγινε η καταστροφή, αλλά φαίνεται από τις στατιστικές ότι εξακολουθούν να πλήττονται από καρκίνο, και ετησίως 21, ε, 21 χώρες ε, υποδέχονται παιδιά από τη Λευκορωσία. Τον Οκτώβριο του 2008 ακούσαμε ότι μέσω διατάγματος της Λευκορωσίας θα απαγορευόταν ε, η... το ταξίδι αυτών των παιδιών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία πλέον να κάνουν το χριστουγεννιάτικο του ταξίδι. Αυτό το διάταγμα περιορίστηκε από 20 Ιανουαρίου έως 20, 20 Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου. Οπότε κάποια παιδιάκια μπόρεσαν να έρθουν στις χώρες μας. Μετά όμως από αυτή την ε, αναστολή δεν ε, μπόρεσαν να συνεχιστούν αυτά τα ταξίδια. Είναι πλέον καιρός να ρυθμιστεί το θέμα αυτό για να μπορέσουν την επόμενη φορά να συνεχίσουν να ταξιδεύουν τα παιδιά αυτά. Εμείς θα θέλαμε να τα ρυθμίσουμε αυτά ε, μία φορά, μία και καλή όχι 27 φορές μέσω σχέσεων. Καλούμε στο ψήφισμά μας την Τσεχική Προεδρία να διαπραγματευτεί με τις αρχές της Λευκορωσίας για μία λύση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μαριάν Μίκο. Ενάμιση λεπτό. Austatud kolleegid, Valgevene tee Euroopasse on dialoogi kompromisside tee Κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη αποτελεί ένα μέρος διαπραγματεύσεων. Πέρσι τονίστηκε η ανάγκη μιας πολιτικής για να υπάρχουν, ε, να τεθούν όροι. Η πρόοδος που σημειώνεται σε διάφορους τομείς αποτελεί πραγματικά προϊόν τέτοια πρόοδου. Ωστόσο, εξακολουθούν να τα προβλήματα που δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Δεν μπορεί τίποτα να, να αντικαταστήσει τη δημοκρατία και ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις καταπιέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών. Δεν μπορεί καμία δημοκρατία να λειτουργήσει χωρίς ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις οργανώσεις που έχουν ως σκόπο την ενίσχυση της δημοκρατίας. Καλωσορίζω την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας για την καταχώρηση του κινήματος για την ελευθερία. Πρόκειται όμως για την αρχή και μόνο. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των σχετικών οργανώσεων. Τέλος, να αναφερθώ στο θέμα των θεωρήσεων. Θα πρέπει να συναυτεί η Συμφωνία Διευκόλυνσης Θεωρήσεων. Ο δρόμος προς την Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Γιατί, αν θέλετε, οι αυστηροί κανόνες για τις θεωρήσεις δεν τιμωρούν την κυβέρνηση, αλλά τον κόσμο της Λευκορωσίας να καλωσορίσουμε τους Λευκορώσους ως Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωκοινοβούλιο δεν ασχολείται για πρώτη φορά με το πρόβλημα της Λευκορωσίας που είναι το ε, τελευταίο δικαθολικό καθεστώ σε ευρωπαϊκό έδαφο. Υπάρχουν δυσκολίες και για τους ε, καθολικούς ιερεί. Δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν αναγνωρίζεται η δημοκρατικά εκλεγμένη οργάνωση των Πολωνών στη Λευκορωσία. Συνεχίζουν οι διώξει σε στα γραφεία των ε, αντικαθεστωτικών, ε, διώκονται οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι κλπ. Πάντως, έστω και με ε, αργά βήματα, γίνονται κάποιες πρόοδοι επιτρέπει καταχώρηση του κίνηματος για την στα Μητρώα, επιτράπει κυκλοφορία δύο ανεξαρτήτων δημοσιο... εφημερίδων κλπ. Και επιτράπει καταχώρηση στα Μητρώα και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βέσνα. Έχουν βελτιωθεί, έχει βελτιωθεί λοιπόν το κλίμα, όπως ανέφερε και η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Μπέρκ για δύο λεπτά. Δεδομένου ότι οι εξωτερικές υποθέσεις είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της ε, Τσεχής Προεδρίας θα μάθω τι πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να, να αρθεί η απαγόρευση ε, μετακίνησης ε, και ταξιδίου των ε, παιδιών από Λευκορωσία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μάθω επίσης τι γίνει με όσους έχουν πληγεί από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Ε, σύμφωνα με την παράφο 10, θα καλούμε το Συμβούλιο της Επιτροπής να εξετάσει τα μέτρα αυτά για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του εμπορίου επενδύσεων κλπ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση Ε, εφάρμοσε μια εξαίρεση που επέτρεπε να ταξιδεύουν τα παιδιά στο εξωτερικό καρδιάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Περίπου χίλιες ε, οικογένειες στην Ιρλανδία ε, φιλοξένησαν παιδιά από την Λευκορωσία και πολλά από αυτά χρειάστηκε να ε, λάβουν και κάποια αγωγή θεραπευτική. Ζητάω λοιπόν από τον Προεδρία να συνεχίσει την πίεση προς την Λευκορωσία έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν τα παιδιά από τη χώρα αυτή να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια απάντηση σε επιστολή μου, κύριε Επίτροπε, είπατε ότι δόθηκαν κάποιες συστάσεις στην Ευρωπαϊκή της στο Μίνσκ. θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ε, έχετε κάποια περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τις ε, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρθεί αυτή η απαγόρευση ταξιδίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, μια βελτίωση των σχέσεων με την Δευκορωσία είναι ε, νομίζω κάτι το οποίο πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Δέχομαι με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δήλωση της Τσεχικής Προεδρίας ε, πάνω στο ζήτημα της ε, συνάντησης την περασμένο μήνα με τους εκπροσώπους της Λευκορωσίας θεωρώ ότι μια τέτοια πρόοδος θα οδηγήσει και σε μια βελτίωση των σχέσεων με τη και την, ότι πρόσφατα με την κρίση του φυσικού αερίου η Δευκορωσία απεδείχθηκε ένας αξιόπτυμος ε, και αξιόπιστος, συγγνώμη, εταίρος. Τη σχέση μας λοιπόν θα πρέπει να τη βασίσουμε στο σεβασμό των δικαιωμάτων και στη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε πέντε άτομα για τη διαδικασία Catch the Η κυρία Πλησίνσκη καταρχάς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Κύριε Βόντρα, ελπίζω να έρθετε πολλές φορές ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακόμα και αν η Λευκορωσία έχει σημειώσει πολλά σημαντικά και θετικά στοιχεία, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με την αντιπολίτευση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη Λευκορωσία. Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να είναι υπό όρου, υπό συγκεκριμένου όρου. Μία, ένας εκ των οποίων θα πρέπει να είναι η ελευθεροτυπία. Τα μέσα μαζική ενημέρωση θα πρέπει να έχουν ελευθερία να λειτουργούν ελεύθερα στη χώρα. Επίση, τα πολιτικά κόμματα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει να έχουν ελευθερία λειτουργία. γιατί πρόκειται για το κλειδί τη δημοκρατία. Όλοι μα θέλουμε μια δημοκρατική Λευκορωσία χωρίς το Λουκασέγκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σημαντική ευκαιρία να κερδίσει τη Λευκορωσία, να την ε, πάρει από την επιρροή της Ρωσίας. Ο κύριος Πατηλόκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε μετά από χρόνια δύσκολων και περίπλοκων ε, σχέσεων ξεκινάμε έναν σωστό δρόμο άδεια σε λειτουργία διάφορων εφημερίδων μη φιλοκυβερνητικών, ε, καταχώρηση του κίνημου για ελευθερία στα Μητρό. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρός, μακρύς. Ξεκίνησαν όμως ε, νέες σχέσεις με την, Ρωσία, την Λευκορωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι θλιβερή η περίπτωση της μη χορήγηση ε, θεωρήσεων σε βουλευτές από πλευρά Λευκορωσίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να φροντίσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν να βελτιωθεί η δυνατότητα μετάβασης ε, ταξιδίου ανηλίκων ε, Λευκορώσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο πλήττει τόσο τις οικογένειές τους όσο και τα ίδια τα παιδιά που έχουν τόση ανάγκη από αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ρίτα. Κύριε Βόντρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, χαιρετίζω τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε με προσοχή την κυβέρνηση του Λουκασέγκο, αλλά πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και να δούμε μια μελλοντική Λευκορωσία μετά το Λουκασέγκα με ένα πολύ θετικό μέλλον. Πρέπει να σκεφτούμε και τον πληθυσμό στην Λευκορωσία, όχι μόνο την κυβέρνηση. Έχει δείξει ιστορία όταν διηγούμε μια χώρα στην απομόνωση, αυτό ευνοεί μια δικτατορία. Είναι εις βάρος του πληθυσμού υπάρχει ένα πρόβλημα όταν κανείς δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να κινηθούν, να πάνε να δουλέψουν, να μετακινηθούν άνθρωποι που αναγνωρίζουν και γνωρίζουν τις αξίες μας. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στον κύριο Φιόρε ότι το ότι οι υποψήφοι φαίνονται στην τηλεόραση, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία, αυτό είναι κάτι θετικό. Ευχαριστώ. Κύριε Σεκέρσκι, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, όλοι που βρισκόμαστε εδώ θα θέλαμε η Λευκορωσία να σεβαστεί τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε και του εκφράζεστε. Θέλουν να πάψουν οι διώξεις των πολιτών και των εθνικών μειοτήτων. Ωστόσο, αυτός ο κατάλογος επιθυμιών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εγγύ μέλλον. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε όμως την προαγωγή των, ανθρωπ... των ευρωπαϊκών αξιών μας. Η πολιτική μας έναντι της Λευκορωσίας ήταν μια καταστροφή κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Ας ελπίζουμε ότι αυτή η μεταστροφή της πολιτικής θα σημειώσει επιτυχία. Δεν πρόκειται να είναι εύκολο όμως. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2008 νοθεύτηκαν από τον Λουκασέγκο για τον εκδημοκρατισμό της ε, Λευκορωσίας χρειάζεται ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας μεταξύ των ε, πολιτών της Λευκορωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ίσως για την νεολαία της ε, Λευκορωσίας. Ευχαριστώ. Please. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μπροστά μου τρεις προτάσεις ψηφίσματος Μαΐου, Οκτωβρίου και αρχές Γενάρη. Βλέπουμε μια εξέλιξη όσον αφορά τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Λευκορισία. Εγώ μπορώ να υποστηρίξω οποιοδήποτε ψήφισμα αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο εκδημοκρατισμό. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε για να ε, βοηθήσουμε στο να υπάρξει διαφάνεια, διαφάνεια η οποία είναι σημαντική για την εξέλιξη της Λευκορυσίας. Και εδώ χρειαζόμαστε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την, ε, μια οριμότητα. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες της Λευκορυσίας τη δυνατότητα να έρθουν πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή ε, Επικράτεια, να έρθουν σε επαφή με τις αξίες μας, να δούνε τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι αξίες που υποστηρίζουμε και μετά μια κίνηση που θα μπορούσε να κάνει ο πρόεδρος Λουκασέγκο να γίνει μια ε, χώρα η οποία δεν έχει πολιτικούς κρατουμένους. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να κάνουμε τη σύνοψη της συζήτησης αυτής. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, να προσπαθήσω να συνοψίσω εκ μέρους του Συμβουλίου. Καταρχάς νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Μια ε, συζήτηση ουσίας, η οποία πραγματικά έφερε πολλά νέα στοιχεία στην κοινή μας εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσω ότι εμείς στο Συμβούλιο εκτιμούμε το ενδιαφέρον και το, τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της Λευκορωσίας. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει ιδιαίτερα θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφενός, αλλά αφετέρου να μην χάσουμε και τη στρατηγική μας αυτή προσέγγιση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα, τους Πολωνούς βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. I think we are listening carefully. Νομίζω ότι πραγματικά ακούμε με μεγάλη προσοχή. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τρία στοιχεία ενίτη συμπερασμάτων. Καταρχάς, για τις θεωρήσεις. Πολύ θίξετε το θέμα αυτό, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σημαντικό. Ακόμα και όταν συζητούμε υπό την εθνική μας ιδιότητα και πέρσι ακόμα, αυτό το θέμα ακούγονταν πάντα πολύ. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν το εξή. Θεωρούμε ότι η Λευκορωσία αποτελεί τμήμα της, Ευρω... της Ευρώπης. Και αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που, ε, από τα οποία, στα οποία υπόκεινται οι πολίτες της Λευκορωσίας. Η Τσεχική Προεδρία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν την ευελεξία που έχουν στη διάθεσή τους σε ό,τι αφορά τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Επίσης, η Προεδρία θα συνεχίσει να ζητά πιο συνεκτική εφαρμογή. Αν δεν τηρηθεί η δυναμική ως έχει, έχουν γίνει άλλωστε σημαντικές ε, πρόοδοι από τη Λευκορωσία. σε τελική ανάλυση θα ξεκινήσει και ένας διάλογος για τις θεωρήσεις. Για τα παιδιά του Τσερνομπίλ. Θέμα που αναφέρατε. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Η Προεδρία μας υποστηρίξαμε μάλλον τις κινήσεις της Γαλλικής Προεδρίας για το θέμα αυτό και για το διάβημα που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου του 8. Τελικά ήταν προσωρινή αναστολή του Ευρωπαϊκού του Προεδρικού Διατάγματος 555. Αυτό στο συνδυασμό με τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες συνήφθηκαν μεταξύ Ιρλανδίας και Λευκορωσίας για τα μελλοντικά ταξίδια των παιδιών αυτό αποτέλεσαν μια μεμονωμένη επιτυχία. Καταλαβαίνουμε φυσικά το γενικότερο πρόβλημα κάθε άλλο παρά έχει λυθεί. Κατανοούμε το μέγεθος του προβλήματος και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αν χρειαστεί. Και θα συνεχίσουμε να θίγουμε το θέμα αυτό στις επαφές μας με τις αρχές στο Μίνσκ. Τελευταία παρατήρηση. Τους επόμενους μήνες με την αθεώρηση των κυρώσεων και στα πλαίσια της μελλοντικής ανατολικής ιστορικής σχέσης, η Λευκορωσία θα παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Όπως και το ψήφισμά σας για τη Λευκορωσία που μας κάλεσε να συνεχίσουμε προς τα εμπρός εμείς, και εμείς ελπίζουμε να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Επιτροπός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, η συντηρητική πλειοψηφία έχει την ίδια άποψη με τη δική μας. Δηλαδή, πράγματι δώσαμε τη δυνατότητα στη Λευκορωσία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και δώσαμε δυνατότητα να ενταχθεί στην ε, πρωτοβουλία για την Ανατολική Ευρώπη και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μερικά από τα σημεία που αναφέρονται. Πρώτον, η οικονομική κρίση, η δημοσιονομική κρίση. Η Λευκορωσία αντιμετώπισε μέχρι τώρα ικανοποιητικά την κρίση αυτή λόγω της ε, ελάχιστης ε, εμπλοκής της στην διεθνή οικονομία. Αλλά τώρα, και ο κ. Μπέλντερ το δήλωσε, είτε θα πρέπει να ζητήσει από το Διεθνές Νομισκατομείο για ένα δάνειο 1,5 δις ευρώ, αλλά και να υποτιμήσει το νόμισμά της προκειμένου να απορροφήσει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης. Επειδή η οικονομία της και η βιομηχανία της ε, δεν είναι σωστά διαρθρωμένες, περιμένουμε αρνητικές επιπτώσεις να συνεχίσουν και να έχουν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Έχετε δίκιο λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό, αυτός είναι ένα σημαντικός παράγοντας. Τώρα, για το για τα πυρηνικά εργοστάσια και το θέμα της ασφάλειας και προστασίας. Έχουμε τεχνικό διάλογο σε θέματα ενέργειας με την Λευκορωσία και από ιδιαίτερη σημασία στο να διασφαλίσουμε πως η χώρα αυτή τηρεί τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και προστασίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Λευκορωσία συνεργάζεται πολύ στενά με την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη και παρέχει πληροφορίες ε, στην Κομισιόν για όλες τις ε, διαδικασίες. Να επανέλθω τώρα στο θέμα των ε, προξενικών θεωρήσεων και του κόστους. Γνωρίζετε πως είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις μόλις τα κράτη-μέλη και ακούσαμε και το Συμβούλιο που εξέφρασε αυτή την άποψη ότι δηλαδή προσπαθεί να πείσει όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ε, με αυτήν την, ε, με την θεώρηση, με τις προξενικές θεωρήσεις και το θέμα της ε, επανειδοχής. Θα ήθελα να σας πω ότι κύριε Μιγκαρέλη ότι για τα τέλη των προξενικών θεωρήσεων και για τις θεωρήσεις ε, για τα παιδιά είναι κάτι το οποίο αφορά κάθε κράτος ε, μεμονωμένα. Δεν υπάρχει μια γενική συμφωνία. Αυτή θα πρέπει ενδεχόμενα να τύχει διαπραγματεύσει ε, από την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Έχουν κατατεθεί πέντε σχέδια ψηφίσματος από το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές, τους φιλελευθέρους, τους πρασίνους, την ΟΕΝ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, η συζήτηση ολοκλώνεται στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε τις εργασίες μας με το επόμενο σημείο στην διάταξη, δηλαδή τη δηλώση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 11η Ιουλίου, μέρα μνήμης των θυμάτων της φραγής ε, της Σρεμπρένιτσα. Το λόγο έχει ο Υπουργό Βόντρα ε, για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη Σρεμπρένιτσα. Όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν εφρικτή η σφαγή περισσότερων από 8.000 Βοσνιών σημάδεψε την Βοσνία Ζεγοβένη, την πρώην Γιουκοσλαβία, αλλά και όλη την Ευρώπη. Αναμφίβολα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ε, αγριότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Κοιτώντα αναδρομικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ, πιο πολλά και πολύ νωρίτερα. Ήταν ένα μια αποτυχία της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για κάτι το οποίο μετανιώνουμε. Είναι ηθικό μας καθήκον και πολιτικό μας καθήκον να μην επαναληφθεί ποτέ η Σρεμπρένιτσα. Η δέκατη επέτειος της ε, σφαγής της Σρεμπρένιτσας αποτελεί φόρο τιμής για όσους χάθηκαν και για τις οικογένειές τους.